Και τώρα ερχόμαστε στις τρεις εκθέσεις που έχουμε του κυρίου Γκουαλτιέρη για την παράταση της θητείας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Τι έγινε, έχετε πρόβλημα. Είναι μυστική η ψηφοφορία, συνάδελφοι. Γι' αυτό βλέπετε το μπλε φωτάκι μπροστά σας. Και τώρα κλείνουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προχωράμε στη δεύτερη έκθεση Γκουαλτιέρη. Και πάλι είναι μυστική ψηφοφορία. Άρχεται. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτη έκθεση, Γκουαλτιέρη, είναι πάλι με μυστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Φοντάνα για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Βοσνίας Ερζεγοβίνης και Ευρώπολα. Ποιοι είστε υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση Νεγκρέσκου για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση της από την Ιρλανδία. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Εάν ψηφίσατε όλοι θα κλείσουμε τώρα την ψηφοφορία. Έγκρινεται. Έκθεση σε δύο τμήματα για το ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Αν θέλω να το ελέγξουμε, είναι ο κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Ελέγχουμε λοιπόν. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολο του κατά αποχές εγκρίνεται έγκριση του γενετικά τροποποιημένου του. Ε, τροπολογία 6 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 4. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική Θέλετε να ελέγξουμε την 5. Μάλιστα. Ελέγχουμε για την τροπολογία 5. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Dodge Niedermayer. Α1 τίτλο Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε Ψηφίζουμε παρακαλώ για την τροπολογία 15. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται Τροπολογία 16 υπέρ. Τι θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Μα συνάδελφοι ήταν σαφέ. Εν πάση περιπτώσει, α το ελέγξουμε. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Έγκρινεται όντω. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ τι θέλετε να ελέγξουμε τη 19 μάλιστα άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστική τροπολογία 9 Σφίζουμε. τέλος απορρίπτεται το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές έγκρινεται αρχικό κείμενο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε τέλος απορρίπτεται το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές Πρέπει να ελέγξουμε για το αρχικό κείμενο. Παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δάφιο 4 ε, και 5 με συγχωρείτε, υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ονομαστική κλίση τροπολογία 12. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13, ονομαστική. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της σύστασης C1. Τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, δύο, μονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο D1 τελευταία παραγράφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 με ονομαστική κλίση, άρχεται, τέλος. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 Δ. υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Ζητήθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας Αλφα τι, υπέρ, το πρώτο τμήματος, δε, ε, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μονομαστική κλίση. Το ψήφισμα. Τέλος. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην άδελφη στην έκθεση Μπέλτερ για τις σχέσεις Ένωσης Κίνας. Παράγραφος 36, αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 38, υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο. Νομίζω έχουμε προφορική από τον κύριο κοφερ; παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο μέσο του κειμένου προτείνω να προσθέσουμε μία πρόταση που λέει Καλή παροτρύνει την Κίνα να επανεξετάσει τη θέση της και ζητά από όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένης της Κίνας να σεβαστούν την ενδεχόμενη απόφαση της Άνκλος. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 ε, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας αβ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία We can now close the vote. And that, colleagues, is adopted. Thank you. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής του κυρίου Γερέρο Σαλωμών. Παράγραφος 11, Πρωτοτμήμα υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Υπέρ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο, τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 23 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 34 τέσσερα τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος της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 Εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Έκθεση Μάρτιν. Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Απλώς θέλω να χαιρετήσω την παρουσία εδώ στο ημικύκλιο μιας αντιπροσωπείας των συνδικαλιστών του Χάλβα που μας έρχονται από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βέλγιο. Πριν να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση για την ανάπτυξη των βασικών μεθόδων, ειδικά για το Χάλβα που υπόκειται σε μια άνευ προηγουμένου κρίση, θέλω να χαιρετήσω την παρουσία τους και τους ευχαριστώ για την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Παράγραφος 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Υπό ε, υπότιτλος 3 ε, υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Υποκατηγορία μάλλον 3, το αρχικό κείμενο, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε το τρίτο τμήμα παρακαλώ τρίτο τμήμα της παραγράφου 11 τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται Παράγραφος 11, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13 υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 13 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται, παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Το αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές. Ελέγχουμε την παράγραφο 14 παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17 σε έξι τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα ονομαστική. Τέλος. εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ε, ονομαστική κλίση, τέλος. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα, άρχεται, τέλος. Έκτο τμήμα, ονομαστική κλίση, τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Έξι τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα. Άρχεται, κλείνει, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση. Άρχεται, τέλος, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκτο τμήμα. Ε, ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε γιατί δεν βλέπω όλα τα χέρια. Ψηφίζουμε λοιπόν. εγκρίνεται. Παράγραφος 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 27, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 29, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 ονομαστική κλίση άρχεται πέρας εγκρίνεται εκτιμώντας D ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας ε, η υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική, άρχεται, τέλος. Εγκρίνεται. H, υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για το εκτιμώντας H. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Ε, εκτιμώντας I, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ε, δεύτερο τμήμα ε, με ονομαστική κλίση τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας M, πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση. Τέλος της πληροφορίας. Ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε. Τέλος της φοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, εκτιμώντας όμικρον ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ποιο, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Εκτιμώντα, ε, τροπολογία 1, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Άρχεται. Είναι ανοιχτή ακόμα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. We now move, colleagues, to the situation... Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Πρόταση ψηφίσματος του ΕΛΚΙΠΕΡ, παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε, να είναι άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Και όντως απορρίπτεται. Περνάμε στην κοινή πρόταση ψηφίσματο τεσσάρων πολιτικών ομάδων, παράγραφος 3, ονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, με ονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7, με ονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη H σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα Μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ, κατά. Αποχές, θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν ε, μπορούν να αποχωρήσουν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ε, πρόταση ψηφίσματος ε, σχετικά με την έγκριση του Γενικού